πρέπει να τα λέμε και πρέπει να τα μεταφράζουμε και σε συγκεκριμένες πράξεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Υπευλήθη από την Επιτροπή την Οικονομική και Νομισματική την Νομισματική Επιτροπή ένα κείμενο ε, Β70318-2010. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο. Εδώ ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι η κοινή συζήτηση για πολιτικές αποδοχών. Έχουμε δύο εκθέσεις της κυρίας Μακάρθη, κεφαλαϊκές απαιτήσει για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για τις θέσεις τιτλοποίησης και νέα τιτλοποίηση για την προληπτική εποπτεία των αποδοχών και η έκθεση του κυρίου Καντράουι καθεστώς αποδοχών των διοικητικών στελεχών των εισηγμένων εταιριών και πολιτικές σχετικά με τις αποδοχές στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Οι δύο εισηγητές θα λάβουν πρώτη το λόγο και πρώτη είναι η κυρία Μακάρθη. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω όλους βοήθ, όσους βοήθησαν για τη Συμφωνία CRD3 για τις κεφαλαιοχικές ανάγκες των τραπεζών. Να ευχαριστήσω την Επιτροπή ΕΚΟΝ και τον προσωπικό και τον Επίτροπο Μπαρνιέ για τη συνεχιζόμενη υποστήριξή του στις προτάσεις της Επιτροπής μας και να ευχαριστήσω και την Ισπανική Προεδρία για την επιμονή και προσπάθειές της σε 12 ωρών τριμερή διάλογο με την διαπραγματευτική ομάδα και τα 27 κράτη-μέλη. Συζητούμε σήμερα για την εφαρμογή των κανόνων της Βασιλείας ε, και ε, τους κανόνες αποδοχών μεταξύ των, που συμφωνήθηκαν από την G20. Όλοι συμφωνούν ότι ο ε, υψηλός κίνδυνος είναι πολύ σημαντικό, σημαντική συνιστόσα που οδήγησε στην κρίση. μετά σε ολόκληρη την Ένωση 3,93 ευρώ δόθηκαν για διάσωση στις τράπεζες. Στο Ηνωμένο Βασίλειο 2,23 ε, ε, δόθηκαν ε, για ένα, που είναι περίπου το ίδιο με ενός έτους ΑΕΠ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ε, οι τραπεζίτες ε, έφυγαν από ε, σόι ενώ μειώθηκαν συντάξεις κλπ. Ο νέος νόμος αντιμετωπίζει αυτά τα βασικά προβλήματα και αδυναμίες στο τραπεζικό σύστημα που οδήγησε στην κρίση. Θα αναγκάσει τις τράπεζες να έχουν μεγαλύτερο κεφάλαιο στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών απέναντι σε κινδύνους. Επίσης θα επηρεάσει τις πρακτικές μπόνους σπάζοντας ε, την ε, ε, αλυσίδα που ενώνει την ανάληψη υπερβολικού κινδύνου και την οικονομική αποζημίωση και επιβράβευση. Είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε την υγεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Αναφέρουν οι τράπεζες ότι έμαθαν το μάθημά τους γιατί η έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας λέει τον Ιούνιο ότι οι αποδοχές, μισθοί και αποδοχές αυξήθηκαν μετά την τραπεζική κρίση και τα 10 δις που κατέβαλαν ε, σε μισθούς και μπόνους ε, στην Αγγλία οι τράπεζες ε, είναι χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να στηρίξουν το κεφάλαιο των τραπεζών και να ε, ε, αυξηθεί το ποσό που διατίθεται στις ε, πιστώσεις στα μικρά νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το οποίο από ό,τι φαίνεται τους τελευταίους μήνες μειώθηκε και η δανειοδότηση θα μειωθεί ακόμη περισσότερο τους επόμενους μήνες. Ε, οι κυβερνήσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση κάνουν περικοπές, ε, μειώνουν τον δημόσιο τομέα, αλλά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με μια τραπεζική κουλτούρα η οποία δίνει, δίνει προτεραιότητα στις αποδοχές των, ε, των στελεχών των τραπεζών. Αυτό επηρεάζει την οικονομική ανάπτυξη. Είναι σημαντικό λοιπόν το 2011 να ισχύσουν κανόνες ε, οι οποίοι ε, προβλέπουν ε, επιστροφή του μπόνους, σύνδεση με το βασικό μισθό, μετοχές, αυξημένη διαφάνεια, βελτίωση της διακυβέρνησης, ούτως ώστε ένας τραπεζίτης ο οποίος είναι υπεύθυνο για τα σφάλματα της τράπεζας του δεν μπορεί να έχει 16 εκατομμύρια φάπαξ φεύγοντας. Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι το, η καταβολή σε μετρητά του μπόνους να είναι περιορισμένο. Ε, η καταβολή ε, μεγάλου μέρους ε, μετρητών, ο, πιστεύει, όπως πιστεύει το Κοινοβούλιο, αποτελεί ένα κίνητρο απαράδεκτο για την ανάληψη υπερβολικού κινδύνου. Ε, ως νομοθέτες έχουμε καθήκον να προασπίσουμε τα συμφέροντα των καταναλωτών και φορολογουμένων. Οι εκλογείς μας θέλουν να δώσουν προτεραιότητα οι τράπεζες στη σταθερότητα και αυτό να ισχύσει και στις αποδοχές και στα μπόνους. Από το 2008 δεν ε, ε, έγιναν μεταρρυθμίσεις. Ε, οι τράπεζες αγνόησαν αυτή την ανάγκη και πρέπει να τους πιέσουμε ούτως ώστε να υπάρχει εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο Ελ Καντράουι έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επιτροπέ, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις ηγητέ για την αγαστή συνεργασία που είχαμε μεταξύ μα. και χάρη σε αυτήν κατορθώσαμε να θεσπίσουμε ένα πολύ συγκροτημένο πακέτο. Η χρηματοπιστωτική κρίση μα έδειξε ότι η πολιτική αποδοχών των υψηλόβαθων στελεχών των τραπεζών στηριζόταν σε μια κοντόφθαλμη προοπτική με ολέθριες συνέπειες για την πραγματική οικονομία, όπως φάνηκε μετά την τραπεζική κρίση. Φάνηκε επίσης ότι οι προαιρετικές συστάσεις έχουν πολύ περιορισμένο αποτέλεσμα. Εμεί θα πρέπει να θεσπίσουμε του κανόνε του παιχνιδιού για να εξασφαλίσουμε η φόρο ανάπτυξη και των εταιριών και τη οικονομία. Η πολιτική συμφωνία για τι κεφαλαϊκέ απαιτήσει που μα παρουσίασε η κυρία Μακάρθη είναι σημαντικό βήμα πρόοδου γιατί αφορά και τη δομή και το μηχανισμό αποδοχών στο χρηματοπιστωτικό κλάδο και ιδιαίτερα την περίπτωση του περιορισμού των επιδομάτων σε περίπτωση κακών επιδόσεων ή της αναστολής και μάλιστα με περίοδο αναφοράς πολυετή. Βέβαια, εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά τα μέτρα δεν είναι επαρκή. Θα πρέπει να θετήσουμε μια ευρύτερη προοπτική και να ενισχύσουμε τους κανόνες της εταιρική διακυβέρνησης, ώστε να ισχύσουν οι ίδιοι κανόνες του παιχνιδιού και εσωτερικέ διαδικασίες στο χρηματοπιστωτικό κλάδο και ε, να ισχύουν παρόμοιες για τις ε, εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες διατάξεις. Επίσης υπάρχουν τα θέματα εσωτερικής και εξωτερικής εποπτείας της πολιτικής αποδοχών των τραπεζών. Συστήνεται η σύσταση μιας ε, ανεξάρτητης επιτροπής αποδοχών που θα είναι υπόλογη προς τους μετόχους και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η μέτοχη του Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές. Επίσης προβλέπεται και μία Επιτροπή Ελέγχου των Κινδύνων ανάλογα με το πακέτο των αποδοχών. Όσοι ασχολούνται με το κίνδυνο θα πρέπει να είναι ανεξάρτητοι με την εταιρεία. Θα πρέπει οι ελεγκτές να μην έχουν συμφέροντα στην εταιρεία για να μπορούν να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα. Και οι συμφωνίες για τη διαχείριση του κινδύνου θα πρέπει να εξετάζονται διεξοδικά από το Εποπτικό Συμβούλιο, ενώ οι εταιρείε θα πρέπει να εφαρμόζουν μια εσωτερική διαιτησία εφόσον υπάρχει διαφορά απόψεων, διάσταση απόψεων μεταξύ του Οπτικού Συμβουλίου και του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίση, οι πρόσθετε αμοιβέ, αυτά τα μπόνου, δεν θα πρέπει να είναι εγγυημένα επαόριστο, θα πρέπει να ανταποκρίνονται στι επιδόσει και στην κατάσταση τη εταιρεία ή τη τράπεζα. Δεν μπορούμε να λαμβάνουμε μέτρα μόνο ποσοτικά, θα πρέπει να θετήσουμε και ποιοτικά μέτρα. Επίσης θα πρέπει να δούμε πόσες, τι διαφορές υπάρχουν μεταξύ των υψηλότερων και των χαμηλότερων αποδοχών. Δεν θα πρέπει να είναι φύρωτα αυτά τα χάσματα. Επίσης θα πρέπει ε, ο υπολογισμός να γίνεται σε ευρύτερη περίοδο και τουλάχιστον το 50% των συμπληρωματικών αποδοχών να δίνονται σε μετοχές. Επίσης θα πρέπει να προβλεφθεί και ένα ανώτατο όριο για τα μπόνους αυτά και τις πρόσθετες αμοιβέ. Δεν θα πρέπει να ξεπερνάει ένα τέτοιο μπόνους ε, το, τις ε, ετήσιες αποδοχές ή τις αποδοχές στο πολύ δύο ετών. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη σύνταξη και τις επικουρικές συντάξεις, θα πρέπει και αυτές να υπολογίζονται με βάση τις επιδόσεις μιας εταιρείας. Επίσης, θα πρέπει να δημοσιεύονται οι αποδοχές όσων υπερβαίνουν το μισό εκατομμύριο ευρώ και να υπάρχει διαφάνεια σε ό,τι αφορά τι συνταξιδοτικέ εισφορέ. Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διερευνήσει, να διερευνήσει έρευνα στα θέματα αυτά και να θεσπίσει και επιπλέον αρχέ πέραν αυτό το πακέτο που έχουμε ήδη εγκρίνει. Για τι συγμένε εταιρείε θέλουμε ένα σύστημα που θα μα δίνει πληροφορίε για το ποιε εταιρείε σέβονται τι συμφωνίε αυτέ και ποιε όχι. Επίση, ε, κύριε Επίτροπε, Περιμένω τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την πράσινη βίβλο για την εταιρική διακυβέρνηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η Κομισιόν έχει το λόγο. Παρακαλώ κύριε Επίτροπε Μπαρινιέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, συζητούμε τώρα μία άλλη πτυχή της απάντησης στην κρίση και των διδαγμάτων που αντλήσαμε από την κρίση μετά την εποπτεία, πώς θα αναμορφώσουμε τις πρακτικές των αποδοχών για να μην ενθαρρύνουμε την ανάληψη υπερβολικών κινδύνων και για το σημείο αυτό και σε σχέση και με τους ίδιους πόρους θέλω να συγχαρώ ε, τους δύο εισηγητές ε, Μακάρθ και Αλκαντράουι τους ε, συνεργάτες τους ε, και τους και όλους εισηγητές ε, που συνεργάστηκαν μαζί τους και όλοι αυτοί δείχνουν πραγματικά πόσο είναι δεσμευμένο το Κοινοβούλιο ε, σε μια πιο σταθερή, πιο υγιή λειτουργία των αγορών ε, που όπως είχα πει και πριν θα πρέπει να υπηρετούν τους πολίτες και όχι να συμβαίνει το αντίστροφο. Αυτό ε, διέπει ε, το έργο της Επιτροπής και του υποφαινομένου κυρίως. Πάντοτε έχω εκφραστεί υπέρ ε, υπεύθυνων επιχειρήσεων ε, που θα είναι στραμμένε προ τον πολίτη, που θα σέβονται την αρχή τη διακυβέρνηση ε, στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και χαιρετίζω τη στήριξη που παρέχει το Κοινοβούλιο σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτό το έργο που έχουμε να επιτελέσουμε. Συμφωνώ με τη διαπίστωση του κυρίου Ελχαντράου. Πράγματι χρειάζονται δεσμευτικά μέτρα για τι πολιτικέ αποδοχών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και με ικανοποίηση ιδιαίτερα η συμβιβαστική πρόταση των τριών θεσμικών οργάνων για την αναθεώρηση των, ε, της οδηγίας ε, για το CRD3 όπως το λέμε που είναι πραγματικά πολύ επικοδομητικές αυτές οι προτάσεις και δίνουν ένα ισχυρό μήνυμα τόσο προς το κοινό όσο ε, και προς τις τράπεζες. Προβλέπεται λοιπόν μεγαλύτερη ρύθμιση, θα υπάρχουν απαιτήσει ιδίων πόρων λοιπόν σε τομείς όπου υπάρχει υποκεφαλαιοποίηση κινδύνων και θα αποφευχθούν πρακτικές ε, πρόσθετων αμοιβών ε, που ενθαρρύνουν την ανάληψη υπερβολικών κινδύνων και που πολύ σωστά έχει καταδικάσει ο Ευρωπαίος πολίτης. Είναι μια σημαντική μεταρρύθμιση που έχει ως στόχο επιτυχές που συνέβαλαν τα μάλα στην πρόσφατη κρίση, το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, ε, οι πολύπλοκες διαδικασίες ε, τιτλοποίησης και οι αποδοχές. Όλα αυτά, ε, όλες αυτές οι προτάσεις και μεταφράζουν στην πράξη τις αρχές του Φόρουμ Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που εγκρίθηκε από την G20 αλλά συγχρόνως βάζουν και αυστηρά όρια ε, στην καταβολή μεταβλητών αποδοχών, αφήνοντας βέβαια και κάποια περιθώρια ελιγμών ε, στις, ε, στους πιστοτικούς οργανισμούς για, σε ό,τι αφορά δε τις αποδοχές, σε ό,τι αφορά τα μπόνους θα είναι περιορισμένα. υπάρχουν σωστοί μηχανισμοί όπως ο μηχανισμός clawback για την επιστροφή αποδοχών σε περίπτωση ανεπαρκούς απόδοσης από 1η Ιανουαρίου 2011 θα ισχύσουν αυτά. Είναι πολύ καλό ε, και σε ό,τι αφορά ε, τα μπόνους που δεν θα έχουν καταβληθεί ακόμη από το 2011, νομίζω ότι θα πρέπει να καλύπτονται από τους νέους κανόνες. Τέλος, προτείνουμε αντίστοιχους κανόνες, ε, κύριοι συγητές και κύριοι βουλευτές, και για άλλους τομείς, όπως είναι οι ασφάλειες, ή τα επενδυτικά ταμεία. Πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη και σεβόμενοι τις ιδιαιτερότητες του κάθε τομέα. Δύο λόγια για την ε, διακυβέρνηση των επιχειρήσεων εν γέννη. Διότι πέρα από τις πτυχές αυτές η έκθεση του κυρίου Λικαντράουι νομίζω ότι απεικονίζει με πολύ εύκολο τρόπο την ανάγκη διακυβέρνηση σε όλε όλες, τι επιχειρήσει. Είναι μια πολύ σημαντική πτυχή για ένα ε, πιο σταθερό ε, ρυθμιστικό πλαίσιο. Έχω ξεκινήσει τι σχετικέ εργασίε. Προτείνω ένα συνολικό θεματολόγιο. Ε, η πράσινη βίβλο τη Δευτέρα είναι του 2010 για την διακυβέρνηση επιχειρήσεων και χρηματοπιστωτικών ευρημάτων είναι ένα πρώτο βήμα προ αυτή την κατεύθυνση. Θα εξετάσουμε τον ρόλο των ελεκτών, των μελών διοικητικών συμβολή συμβουλίων όλων όσων έχουν κάποια ευθύνη ή αρμοδιότητα. Αυτά άλλωστε τα ζητά και η έκθεση του κ. Λικαντράουι η οποία επίσης ε, αναφέρεται και σε θέματα σύγκρουσης συμφερόντων ε, στο ρόλο και στη λειτουργία ε, της διοικητικής διαδικασίας, διαχείριση κινδύνων, ρόλος μετόχων, εποπτών και ελεγκτών στα διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Για αυτούς τους δύο μήνες που ακολουθούν θα έχουμε σημαντικές διαβουλεύσεις. Και επαναλαμβάνω, θα έχουμε επέκταση της διακυβέρνησης ε, και σε άλλους τομείς όπως διαφοροποίηση, θέση γυναικών ε, στην, ε, και εκπροσώπησή του στα διοικητικά συμβούλια και ούτω καθεξής. Ένα τρίτο θέμα είναι ο εξυγχρονισμός του Ταμείου των Ιδίων Πόρων. Ρύθμιση είναι μια πτυχή πέραν των ιδίων πόρων κινδύνου σε περίπτωση τραπεζών που προκαλούν κρίση ξέρουμε ότι δεν επαρκούσαν τα μέτρα τα οποία είχαμε μέχρι τώρα για την κράτηση κεφαλαίου. Θέλουμε να ενισχύσουμε λοιπόν τη ρύθμιση, να διορθώσουμε κάποια κενά σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο που σχετίζεται με το, και τον υπολογισμό του που σχετίζεται με το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και να έχουμε και ένα επαρκέ επίπεδο ε, διακρατηθέντο ε, κεφαλαίου. Ίσως κάποιοι φοβάστε ότι δεν θα εφαρμοστούν ε, μέχρι τα τέλη του 2011 οι πολύ σημαντικέ αυτέ μεταρρυθμίσει ε, και εγώ έχω υπόψη μου τον κίνδυνο αυτό. Όταν, παραδείγματο χάρη, φάνηκε ότι στη ΣΥΠΑ δεν θα μπορούσαν οι νέοι κανόνε Επιτροπή Βασιλεία να εφαρμοστούν πριν τα τέλη του 2010, εγώ στην πρόσφατη επίσκεψή μου στη ΣΥΠΑ το επισήμανα ε, στον αρμόδιο υπουργό, τον Τίμωθη Γκάρτνερ και Συμφωνήσαμε να υπάρξει ημερομηνία για την εφαρμογή αυτών των νέων κανόνων. Το Μάιο συγκεκριμένα συμφωνήσαμε. Η Επιτροπή της Βασιλείας ε, λοιπόν, ε, κατέληξε στο ότι πριν το τέλο του 2011 θα έχουν εφαρμοστεί αυτοί οι νέοι κανόνε. Πρόκειται για μια ευέλικτη παγκοσμιοποιημένη αγορά. Αυτή η σύγκληση και ιδίω μεταξύ Ευρώπη και Αμερικής είναι πάρα πολύ σημαντική. Νομίζω ότι διαπραγματευόμενοι την προθεσμία αυτή έχουμε εξασφαλίσει με μεγαλύτερη βεβαιότητα ότι όλοι οι διεθνεί εταίροι μεταξύ αυτών και πρώτα απ' όλα οι Αμερικανοί εταίροι μα θα εφαρμόσουν τους ε, κανόνε αυτού με βάση το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα. Πιστεύω ότι ε, πρέπει να πούμε ότι κάποιες φορές ήταν δύσκολες, πολύ δύσκολες οι διαπραγματεύσεις. Θέλω να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά την, Αλέν, ε, την Αρλέν Μακάρθη και τους ε, σκιώδεις εισηγητές για την προσπάθειά τους, για την διαθεσιμότητα και ήμουν ε, ιδιαίτερο ευτυχής που και εγώ και οι συνεργάτες μου συνεργαστήκαμε μαζί σας. Και τώρα ο κύριος για την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα οικονομικά κίνητρα, οι αποδοχές, τα μπόνους είναι γνωστά στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Και μεταξύ άλλων και αυτές οι αποδοχές και τα κίνητρα και πόνου συνέβαλαν στη χρηματοπιστωτική κρίση. Γι' αυτό θα πρέπει να τροποποιήσουμε την οδηγία και να την προσαρμόσουμε στις νέες ανάγκες και εξελίξεις. Θα ήθελα να συγχαρώ τους ηγητέ για το έργο τους. Στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων εξετάσαμε αυτό το θέμα τη πολιτική αποδοχών και χαιρόμαστε για τις παραγράφους που ζητούν διαφάνεια και καλή ενημέρωση όλων των εταίρων των μετόχων, δηλαδή των αρμόδιων αρχών, των μισθωτών και ούτω καθεξής. Σχεδόν ομόφωνα η Επιτροπή Απασχόλησης τάχθηκε κατά των options. Πρόκειται για ορισμένα κίνητρα που οδήγησαν ουσιαστικά στην ανάληψη των κινδύνων και το πρόβλημα αυτό είναι γνωστό. Ακόμη και ο χρηματοπιστωτικός κλάδος γνωρίζει αυτά τα θέματα. Είμαστε κατά οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων, ο κυρίος Σότμαρ Κάρας, 1,5 λεπτό εξ ονόματος του ΕΛΚΕ. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, άρχισαν να κινούνται πάλι ε, τα πράγματα στο Συμβούλιο και αυτό είναι ένα πολιτικό μήνυμα. Δεν ξέρω αν ε, έχουν όλοι επίγνωση ε, αυτής της εξέλιξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, τάσεται υπέρ σαφέστερων κανόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θέλουμε ανώτατα όρια, θέλουμε ε, δυνατότητες πληρωμών που μειώνουν το κίνδυνο. Είμαστε υπέρ της ανάληψης ευθύνης των περιορισμών των πόνους ε, των τραπεζικών στελεχών με τα ε, μετρητά να μην είναι υψηλότερα από το κεφάλαιο επίσης, το, ε, που διατίθεται για τους κινδύνους. Ε, είναι πολύ σημαντική η συμφωνία του Επιτρόπου Μπαρνιέ με τους Αμερικανούς σε σχέση με το χαρτοφυλάκιο των τραπεζών και το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών. Είναι σημαντικό να γίνει η προσαρμογή αυτή των χαρτοφυλακίων. Επίσης ενισχύθηκαν οι κανόνες γνωστοποίησης, η ε, εναρμόνιση του κινδύνου στα δύο χαρτοφυλάκια και είναι πολύ σημαντικό να ε, υπάρχουν διαθέσιμα για περιόδους κρίσης χρειάζεται επίσης να, ε, ε, η ενίσχυση και οι αυστηρότεροι κανόνες για το χαρτοφυλάκιο των συναλλαγών. Θα πρέπει να ξεπεράσουμε το πρόβλημα των ε, πτωχεύσεων. Θα πρέπει να δράσουμε πολύ περισσότερο προληπτικά. Εξ ονόματα σοσιαλιστών και δημοκρατών, ο κύριος Λούντβιχσον για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα αυτό προκάλεσε σφοδρές συζητήσεις τα τελευταία χρόνια. Το θέμα της πολιτικής αποδοχών και των πόνους των στελεχών ε, των τραπεζών. Μέχρι στιγμής ε, είχαμε μάλλον αδύναμα μέτρα και νομοθεσία. Τώρα χρειαζόμαστε μια πιο στεναρή νομοθεσία που ελπίζουμε ότι θα μειώσει την ανάληψη υπερβολικού και του κινδύνου. Και στο μέτρο που ο κίνδυνος ε, θα περιοριστεί, η σταθερότητα θα ενισχυθεί. Ο χρηματοπιστωτικός κλάδος θα έπρεπε εδώ και πολύ καιρό να ε, βγάλει αυτά τα επικίνδυνα συστήματα των πόνους ε, και επιδοτήσεων υπερβολικών αποδοχών και δυστυχώς δεν το έκανε. Είναι σημαντικός ο κίνδυνος για την κοινωνία να δεχτούμε μια τέτοια κατάσταση αδιαμαρτύρητα. Οι φορολογούμενοι έχουν πληρώσει τα σπασμένα και έχουν σώσει τις τράπεζες, έχουν καλύψει τα ελλείμματα των τραπεζών. Ελπίζουμε η οδηγία αυτή να εφαρμοστεί από τα κράτη-μέλη το συντομότερο δυνατό προκειμένου να ισχύσουν παντού οι κανόνες. Ευχαριστώ. Και τώρα εξ ονόματος ε, των ε, φιλελεύθερων δημοκρατών, η κυρία Μπόλς, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Ε, κύριε Επίτροπε, η μεταρρύθμιση σε αυτό το τομέα είναι το πιο σοβαρό νομισματικό, ε, νομοθετικό μέτρο μετά την κρίση και ε, χρειάζεται να προχωρήσουμε πέρα από το, την αρχιτεκτονική εποπτείας. Είναι σημαντικά τα μπόνους για την κρίση ε, και δημιούργησαν μια φιλοσοφία υπέρ του κινδύνου και τις ρηψοκίνδυνες ενέργειες. Θα πρέπει λοιπόν αυτά τα συναλλακτικά ήθη να τροποποιηθούν. Ε, αυτό είναι πολύ σωστό γιατί πιάνουμε τη ρίζα της κρίσης και του τραπεζικού συστήματος. Για, τους, για τις αποδοχές ε, μεγάλα μπόνους, ε, μεγάλα εφάπαξ. Ε, πολλοί είχαν πει ότι δεν θα πρέπει να τα αλλάξουμε. Είναι πολύ σημαντικό ότι υποστηρίχθηκε αυτή η ιδέα να γίνουν τα κεφάλαια αυτά, κεφάλαια εκτάκτου ανάγκης. Λυπάμαι γιατί δεν μπόρεσε να ενταχθεί και το κείμενό μου σε σχέση με την φοροδιαφυγή. Πάντω νομίζω ότι με τις τροπολογίες ευελτιώνεται η οδηγία. Εξ των Πρασίνων, ο κύριο Κανφέ, δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ. Καλησπέρα κύριε Επίτροπε. Η δική μου πολιτική ομάδα χαίρεται ιδιαίτερα ε, με την έκθεση της οδηγίας αυτής ε, η οποία περιλαμβάνει δύο στοιχεία αποδοχών. Πρόκειται ίσως για τους πιο φιλόδοξους ε, κανόνες στον κόσμο. Η ικανότητα σημαντικού περιορισμού των μεταβλητών αποδοχών των διευθυντών των τραπεζών ή ακόμη και η δυνατότητα αναστολής της καταβολής και του 60% ε, του ποσού για να ληφθούν υπόψη τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της ε, ε, τράπεζας, οι κίνδυνοι και οι, αρνητικοί, οι αρνητικές συνέπειες για να μειωθούν αυτές οι πρόσθετες αμοιβές. Όλοι αυτοί οι κανόνες είναι σημαντικοί που μεταφράζουν σε συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο τις δεσμεύσεις αρχής της ομάδας των 20. Όπως και οι άλλες κοιόδες εισηγητές, με την εισηγήτρια κυρία Μακάρθη, αναφερθήκαμε πολλές φορές στην κακή βούληση των κρατών, στο απίστευτο χάσμα μεταξύ των λόγων για ε, την, ε, τον ανήθικο χαρακτήρα του καπιταλισμού ε, κτλ. αφενός, αλλά την στάση του Συμβουλίου και των σημαντικών κρατών που προσπαθούσαν συνέχεια να καθυστερήσουν, να παρακολύσουν την εκτέλεση των δικών μας φιλόδοξων προτάσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έλεγα ότι μάλλον ήταν περισσότερο στο δικό μας στρατόπεδο και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πολύ θετικό, είναι ένα κεκτημένο που μας χαροποιεί. Τώρα, κάναμε συμβιβασμούς, χάσαμε κάποιες μάχες ε, ε, σε ό,τι αφορά την ποσοτικοποίηση, ε, δηλαδή δεν έχουμε συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία, αλλά έχουμε κάποιες λέξεις, δικαιολόγηση, και εξισορρόπηση κτλ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα θα πρέπει αυτές τις λέξεις να τις, αυτούς, αυτά τα σημεία αναφορά θα πρέπει να τα μεταφράσει σε συγκεκριμένα ε, αριθμητικά στοιχεία. Και θα ήθελα να δω, κύριε Μπαρνίε, πώ εσεί ε, θα ασκήσετε πιέσει και πώ θα εξασφαλίσετε ε, τον έλεγχο, τον αυστηρό έλεγχο τη εφαρμογή τη διαδικασία, ώστε το κείμενο το οποίο θα ψηφίσουμε αύριο να μην αλλοιωθεί και να χάσει την τόλμη του στο πλαίσιο τη μελλοντική διαδικασία. Ο κύριο Όμπερ Μάιερ, μη εγγεγραμμένο. Ευχαριστώ. Μάθαμε από την κρίση γιατί δεν μπορούμε ανεύθυνες ε, πολιτικές να τις συνεχίζουμε. 20%, ε, 30% είπαμε καταβολή σε μετρητά ε, με προϋποθέσεις. Αυτό δίνει μηνύματα και στους φορολογουμένους που εκλήθησαν να πληρώσουν πολλά χρήματα και δεν καταλαβαίνουν γιατί οι ανεύθυνοι μάνατζερ να παίρνουν τέτοια μπόνους. Εδώ πρόκειται για μια πρωτοφανή διεθνώς ρύθμιση, ούτω ώστε να αποφύγουμε προβλήματα με τη Νέα Υόρκη ή το Τόκιο. Θα πρέπει να ε, έχουμε και κοινή ε, ε, ρύθμιση σε περισσότερους τομείς. Πιστεύω ότι θα πρέπει να εμποδίσουμε οδούς διαφυγής για ανεύθυνους ανθρώπους. Επίσης, οι προδιαγραφές για την εταιρική διακυβέρνηση ε, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους και την, τον περιορισμό των αποδοχών και σε μη εταιρείε. Αυτό θα συμβάλλει στην ε, οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση ε, παγκοσμίω. Και τώρα οι, ε, οι υπόλοιποι ομιλητές που έχουν ζητήσει το λόγο, ο κύριος Νίτρας, 1,5 λεπτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, Νομίζω ότι κάναμε ένα πολύ σημαντικό βήμα σήμερα προσπαθώντας να διαθετήσουμε την πολιτική αποδοχών των τραπεζών. Οι αποδοχές, οι αμοιβέ των στελεχών ε, έφτανε, έφταναν στα αστρονομικά ποσά και σε μεγάλο βαθμό οδήγησαν στη χρηματοπιστωτική κρίση. Θα πρέπει λοιπόν από κοινού να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε το ρόλο του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και των εποπτικών αρχών, να ενισχύσουμε και τον εσωτερικό και τον εξωτερικό έλεγχο. Νομίζω ότι καταλήξαμε σε συμφωνία ότι χρειαζόμαστε κάποιες κοινέ ε, διατάξεις, κάποιους κοινού κανόνες. Για παράδειγμα, ζητούμε μια απολύτως ανεξάρτητη εποπτική αρχή. Και είπαν οι προλαλήσαντες ότι ένα σημαντικό τμήμα των πόνους θα πρέπει να συσχετίζονται με τις μακροπρόθεσμες επιδόσεις και τα επιτεύγματα των στελεχών. Κάτι άλλο επίσης είναι πολύ σημαντικό, ότι η πολιτική των αποδοχών, που μέχρι στιγμής ήταν σαφώς εσφαλμένη, δεν ήταν ε, ούτε ο μοναδικός παράγων, ούτε ο κυρίαρχος παράγων της κρίσης. Και αν είχαμε τέτοιους, ε, τέτοια συμπεράσματα θα καταλήγουμε σε ανακριβείς ε, αναλύσεις της κρίσης και δεν νομίζω ότι θα καταφέραμε έτσι να λάβουμε σωστά μέτρα. Σε ευχαριστώ θερμά τους συγητές για τις εκθέσεις τους. Ο κύριος, ε, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Είμαι ο σκιώδης συγητής για τη δεύτερη έκθεση και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή μας, τον κύριο Χαντράουι, για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε κατά την εκπόνηση της έκθεσής του. Φυσικά, δεν ε, μας εξέπληξε η διαπίστωση ότι χρειάζεται κάποια παρέμβαση στον τομέα αυτό. Μερικές φορές βέβαια τα επιχειρήματα υπέρ της παρέμβασης έχουν ε, κάπως δημαγωγικό χαρακτήρα. Θα πρέπει φυσικά να καταλήξουμε σε μια σωστή πολιτική συναλλαγών δεν μπορούμε να συνεχίσουμε την πολιτική των τελευταίων ετών, γιατί αυτή μας δημιούργησε πολύ άριθμα προβλήματα. Ταυτόχρονα θα πρέπει να αποφύγουμε τις ε, άκρητες γενικεύσεις. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι δεν είναι προς το συμφέρον των επιχειρήσεων να συνεχίσουν μια τέτοια πολιτική ιδιαίτερα επικίνδυνη σε θέματα δανείων. δεν θα πρέπει να τα βάζουμε όλα σε δύο τσουβάλι, θα πρέπει να κάνουμε σημαντικές διακρίσεις. Ο κύριος Μπάλτς, μισή λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο Ότμαρ Κάρας, ήδη είπε σημαντικά πράγματα, συμφωνώ απόλυτα. Χρειαζόμαστε ποσοτικά και ποιοτικά καλύτερες προδιαγραφές για κεφαλαιακές ε, ε, στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ε, είναι πολύ ε, σημαντικό να προχωρήσουμε με τρόπο παραγωγικό. Η χρηματοοικονομική κρίση είναι παγκόσμια. Θα πρέπει λοιπόν οι κινήσεις να γίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Εάν κάνουμε αυστηρότερες τις προδιαγραφές για κεφαλαιακή επάρκεια πρέπει να το κάνουμε ε, συντονισμένα. Οι ίσοι όροι του παιχνιδιού πρέπει να ισχύουν και βλέποντας τις αποφάσεις με, για τις συμφωνίες με τους Αμερικανούς φίλους διατηρώ κάποιες αμφιβολίες. Επίσης η ε, δεν πρέπει να, ε, των προγραμμάτων θα πρέπει να γίνει συντονισμένα και εναρμονισμένα. Είναι πολύ σημαντικό ε, να γίνει σωστή ερμηνεία και από την εποπτική αρχή στο μέλλον. Μην ξεχνάμε ότι η πραγματική οικονομία, η χρηματοοικονομική αγορά αλληλοεπηρεάζονται. Μέχρι τώρα δεν ξέρουμε ακριβώς πώς. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε εκτιμήσεις ε, των επιπτώσεων πριν αλλάξουμε το νομικό πλαίσιο. Αυτή ήταν η διαπραγματευτική γραμμή του ΕΛΚ. Ο συμβιβασμό με το Συμβούλιο που εξευρέθη πιστεύω ότι είναι η μόνη λογική λύση και ευχαριστώ πάρα πολύ ε, τους συναδέλφους Μακάρθη και Κάρασε για την εργασία του ε, στα πλαίσια αυτής της ε, έκθεσης. Ευχαριστώ και εσάς. Και τώρα περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye. Πρώτος έχει το λόγο Α, πρώτα η κυρία Αντζελίλη, παρακαλώ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία, κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ θερμά και τους δύο εισηγητές για το καταπληκτικό τους έργο. Η πολιτική αποδοχών και περιορισμό των αποδοχών των ε, σούπερ μάνατζερ είναι πολύ σημαντικό μήνυμα γιατί για πρώτη φορά σε παγκόσμιο επίπεδο προβλέπουμε ένα ανώτατο όριο σε ό,τι αφορά τι αποδοχέ των ε, τραπεζικών στελεχών. Πρόκειται για ένα πακέτο σαφών μέτρων και λέμε ότι οι επιδοτήσεις στα μπόνου των μάνατζερ θα καταβάλλονται εφόσον η τράπεζα εισέπραξε το κέρδο και όχι μόνο επί τη βάση των προβλέψεων των αποτελεσμάτων. Τρίτον, τα νέα μέτρα θα θέσουν επιτέλους τέρμα στην ενθάρρυνση ανάληψη ασυλλόγιστων και υπερβολικών κινδύνων. Αποκαθίσταται μεγαλύτερη διαφάνεια και εμπιστοσύνη και ευθύνη για τους μετόχους που, συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις και ασκούν το δικαίωμα ψήφου τους σε ό,τι αφορά το επίπεδο αποδοχών των ε, διοικητικών στελεχών. Ο κύριος Μικολάση και ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε τα υπερβολικά, ε, οι υπερβολικέ αποδοχές οδήγησαν στην ανάληψη υπερβολικών κινδύνων και αυτό ήταν κάτι πολύ κακό για τους υπαλλήλου, τον χρηματοπιστωτικό τομέα και οικονομίε ολόκληρων χωρών. Και ήταν ένας από τους παράγοντες πίσω από τη χρηματοπιστωτική κρίση. Γι' αυτό χαιρετίζω την πρωτοβουλία ρύθμιση ε, των αποδοχών στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Πολύ συχνά τα ανώτερα στελέχη κινούνται με γνώμονα το προσωπικό όφελο και λαμβάνουν κινδύνου οι οποίοι έρχονται σε αντίθεση με το συμφέρον των μετόχων και του χρηματοπιστωτικού ιδρύματο στο οποίο εργάζονται. Ιδίω όταν οι φορολογούμενοι είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει μετά να σώσουν την κατάσταση και να διασώσουν τα χρηματοπιστωτικά αυτά ιδρύματα. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει υψηλό ποσοστό διαφάνεια στι αποδοχέ. Επιπλέον θα πρέπει οι μέτοχοι να έχουν μεγαλύτερη εξουσία, μεγαλύτερη δύναμη. Δυστυχώ τελείωσε ο χρόνο σα. Ο κύριο Μόλτσερ, ένα λεπτό παρακαλώ. Στην Αυστρία ε, κλείνουν ταχυδρομεία ε, όμως ε, οι αμοιβέ ε, ε, των ανωτέρων στελεχών αυξήθηκαν κατά 40%. Αυτό δεν γίνεται κατανοητό, ούτε μπορούμε εύκολα να βγάλουμε συμπεράσματα. Ο γερμανικός νόμος για την σωστή δομή των αποδοχών δημιούργησε ένα ενδιαφέρον γύρω από το σύστημα των αποδοχών και ε, δημιουργήθηκαν και νέες ε, διασφαλίσεις που όμως δεν απέδωσαν. Αυτό θα πρέπει να οδηγήσει σε κάποια άντληση διδαγμάτων. Ε, είναι σαφές ότι όταν αυξάνονται οι αποδοχές σημαίνει ότι θα πρέπει και η μάχη μας να κλιμακωθεί. Είναι σημαντικό επίσης να υπάρχει ε, διαφάνεια ε, στο σύστημα από το οποίο εξαρτώνται τα μπόνους. Ευχαριστώ. Η κυρία Μαγκίνες, ένα λεπτό πάλι. Ευχαριστώ. κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω του συζητητέ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι εξειδικευμένο το θέμα, αλλά νομίζω ότι όλοι οι πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση χαίρονται που Συμβούλιο, Κοινοβούλιο και Επιτροπή αντιμετωπίζουν το ζήτημα των υπερβολικών αποδοχών. Γνωρίζουμε όλοι τι ε, υπερβολέ οι οποίε προέβησαν κάποια στελέχη τραπεζών λόγω των καταστροφών ε, που βιώσαμε οι αποδοχές πραγματικά έχουν ξεφύγει εντελώς ε, και ε, αυτό το αντιλαμβάνεται η κοινή γνώμη. Πρέπει να πω ότι κλειδίνει η διαφάνεια. Πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος τι συμβαίνει, πρέπει να μπορούμε να αναλάβουμε δράση. Από τους ε, πιο χαμηλός, χαμηλόμιστους κτηνοτρόφους και γεωργούς δημοσιεύονται οι αποδοχές τους, το μισθολογιό τους. Το ίδιο θα πρέπει να γίνεται και για τους τραπεζικούς. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα. Βέβαια, δεν είμαι πεπισμένη σημαίνει ότι η νοοτροπία των τραπεζιτών έχει αλλάξει και θα πρέπει πραγματικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι πολύ αυστηρή γιατί αλλιώς ε, θα γυρίσουμε στην ε, προηγούμενη κατάσταση φοβούμε. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν, ο Επίτροπος Μπαρνιέ. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. με συγκινή εμπιστοσύνη που δείχνετε απέναντί μου, γιατί με τέσσερις ώρες εδώ και παρόλα αυτά δεν έχετε κουραστεί να με ακούτε. Άκουσα και εγώ τις απόψεις στα πολύ σημαντικά αυτά θέματα και ευχαριστώ θερμά την Αριλίν Μακάρθη και τον Σαϊντ Αλκαντράουι καθώς και όλα τα μέλη της Αρμόδιας Επιτροπής για την αφοσίωσή του στην επιμέλεια, τη συμβολή τους ε, στη σημαντική βελτίωση της πρότασης. Κυρία Μακάρθη, βελτιώσετε σημαντικά το κείμενο. Βέβαια, πολύ δρόμο έχουμε ακόμη να διανύσουμε σε αυτό το θέμα του χρηματοπιστωτικού κλάδου και τη πολιτική αποδοχών και σε άλλου χρηματοπιστωτικού τομεί, την διακυβέρνηση, την εταιρική διακυβέρνηση, τα παράγωγα προϊόντα, τις πωλήσει θα προτείνουμε σχετική τροπολο... ρύθμιση ήδη από το Σεπτέμβριο. Επίσης την εγγύηση των καταθέσεων, την αντιστάθμιση των επενδυτών και αναμένεται και μία λευκή βίβλος για τις εγγύησει στον τομέα των ασφαλίσεων. Το κείμενο, τα δύο κείμενα, οι δύο εκθέσεις που θα ψηφίσετε αύριο νομίζω ότι είναι πολύ καλές. Και ενσωμάτωσαν πολλές τροπολογίες στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων χάρη στην συνεισφορά της Επιτροπής σας. Για παράδειγμα, λεπτομέρειε ότι αφορά τον υπολογισμό των αποδοχών και τη διαφάνεια τη πολιτική αποδοχών ή κάποιου περιορισμού ε, των πόνου ε, κάποιων ε, τραπεζικών ιδρυμάτων που έλαβαν κρατικέ ενισχύσει και το θέμα του Clawbank, τη δυνατότητα αναστολή των πόνου. Επίσης, η αρχή του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για τι αποδοχέ είναι πολύ σημαντικό θέμα. Και υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των κρατών μελών σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό. Εξού και οι γενικές αρχές του Χρηματοπιστωτικού Συμβουλίου αφήνουν μεγάλο περιθώριο ελιγμό στα κράτη-μέλη, αλλά θα πρέπει να εφαρμόσουμε μια συνεπή εφαρμογή της, της οδηγίας από τα κράτη-μέλη. Χρειαζόμαστε σαφείς κανόνες και όχι αποκλίνουσες ερμηνείες. Θα πρέπει να τονίσουμε αυτή την ανάγκη ε, συνεκτικής ε, και συνεπούς εφαρμογής της οδηγίας για να μην αφισβητηθεί εξαιτία της ε, διαφορετικής εφαρμογής της οδηγίας η ανταγωνιστικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλωστε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πρώτη ήπειρος που προβλέπει τέτοιες ρυθμίσεις και προτάσεις για ευφύ διακυβέρνηση των τραπεζών. Έχουμε βέβαια και νέες ευρωπαϊκές αρχές συνεχίζονται για το θέμα αυτό οι διαπραγματεύσει στο Συμβούλιο. Οι νέε αυτέ αρχέ θα πρέπει να έχουν ένα γνήσιο, μια γνήσια εξουσία συντονισμού και αρμοδιότητα συντονισμού και να συμβάλλουν στην συντονισμένη και συνεκτική εφαρμογή των κοινών κανόνων. Και επίση να λαμβάνουμε μέτρα σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται σωστά το κοινοτικό δίκαιο, ακόμη και σε ό,τι αφορά του κανόνε για τι αποδοχέ. Θα είμαστε ιδιαίτερα ιδιαίτερα προσεκτική στα θέματα αυτά. Οι νέοι κανόνε θα πρέπει να εφαρμόζονται από όλε τι τράπεζε, από τα επενδυτικά όργανα επίση και φορεί και προβλέπουμε ε, κάποιε αρχέ αναλογικότητα ώστε να εφαρμοστούν από τα διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ανάλογα με το μέγεθό του, ε, τη νομική του δομή, την πολυπλοκότητα τη φύση του και το είδο των δραστηριοτήτων του χάρη στη συμβολή σας ε, θα αλλάξουν σημαντικά οι πρακτικές που πολύ συχνά ίσχυσαν μέχρι τώρα και που συνέβαλαν στην ανάληψη υπερβολικού κινδύνου από πλευράς τραπεζών και μας οδήγησαν στη σημερινή χρηματοπιστωτική κρίση. Ευχαριστούμε κύριε Κάρας για την υποστήριξή σας ότι αφορά την εφαρμογή αυτών των μέτρων παράλληλα με τις ΗΠΑ. Ό,τι αφορά το θέμα του δικαίου αφαιρεγκαιότητας θα το εξετάσουμε στα πλαίσια του προγράμματος για την ε, επίλυση των κρίσεων. Αλλά αυτό είναι πιο μακροπρόθεσμο και μακρόπνο σχέδιο. Αναφέρθηκε το θέμα της διαφάνειας. Είναι πολύ σημαντική η διαφάνεια και είναι ένα θέμα για το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέμενε και βελτίωσε πολύ σημαντικά τις αρχικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η κυρία Μπόλς αναφέρθηκε στο μείζον θέμα της κεφαλαιοποίησης και ο κύριος Μπάλτς ε, πριν από λίγο το ίδιο είπε. Φυσικά είναι σημαντική η κεφαλαιοποίηση, αλλά εξίσου σημαντικό είναι ένα καλό πλαίσιο εσωτερικής και εξωτερικής εποπτείας, ένα θέμα που θα μας απασχολήσει σε άλλη περίπτωση. Φυσικά η Συμφωνία της Βασιλείας θα είναι πλαίσιο και σίγουρα θα ληφθούν υπόψη και οι μελέτες επιπτώσεων καθώς και μακροοικονομικές μελέτες που θα είναι απαραίτητες ε, για να εξασφαλίσουμε τη σωστή ε, εφαρμογή των μέτρων. Θα πρέπει να δούμε πώς θα συνδυαστούν αυτά τα μέτρα της Βασιλείας με τα άλλα μέτρα της πρόληψης, της προφύλαξης, εσωτερικής και εξωτερικής εποπτείας, ε, επίλυση των διαφορών, ο μηχανισμό της εποπτείας και επίσης ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα είναι να δούμε τι κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες από τη μια πλευρά και τι θα κάνουμε εμείς στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Φυσικά ε, το G20 έθεσε κάποιους στόχους και πιστεύω ότι θα πρέπει και εμείς, ε, εκ με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να φροντίσουμε και την υλοποίηση αυτών των στόχων. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Οι η κυρία Μακάρθη Πολύ σύντομα συμφωνώ ότι δεν άλλαξε η νοοτροπία και η κουλτούρα και μάλιστα τελευταία ε, κάποιες τράπεζες ε, προσπάθησαν να υπονομεύσουν τις προτάσεις που θα ψηφίσουμε αύριο Γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουν οι ρυθμιστικοί φορείς ως θένος να υπερασπιστούν την ε, νομοθεσία, να δώσουμε ένα ισχυρό μήνυμα στο, στην κοινή γνώμη ότι θέλουμε να κάνουμε τη μεταρρύθμιση αυτή, να μετασχηματίσουμε το, την κουλτούρα του μπόνους. Είναι η αρχή της διαδικασίας, όχι το τέλος. Γι' αυτό ε, θα ήθελα να παρακαλέσω τους συναδέλφους αύριο στην Ολομέλεια να υπερψηφίσουν την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Κύριος ε, Ελκαντράουι, δύο λεπτά. Ε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα είμαι σύντομος. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι χρειάζονται νέοι κανόνες για την πολιτική αποδοχών και είναι επίσης σαφές και το δείχνουν και οι εξελίξεις των συστάσεων της Κομισιόν ε, μετά από την πρώτη πριν από ένα χρόνο για τις αποδοχές ότι θα πρέπει οι συστάσεις αυτές να είναι όσο γίνεται πιο δεσμευτικές. Βέβαια δεν είναι όλοι πρόθυμοι να προχωρήσουν ως το ίδιο σημείο, δεν έχουν όλοι τις ίδιες φιλοδοξίες. Θα πρέπει όμως να συμφωνήσουμε όλοι ότι αυτά που συζητούμε σήμερα και που ελπίζω αύριο θα εγκρίνουμε αποτελούν ένα πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν μπορεί όμως να είναι το τελευταίο βήμα. Ακόμα μένει πολλή δουλειά να γίνει θα πρέπει και ο εξωτερικός έλεγχος της πολιτικής αποδοχών στις επιχειρήσεις να ενισχυθεί. Ο ρόλο των επιτροπών αποδοχών πρέπει να διευκρινιστεί. Επίσης η σύνδεση με τη διαχείριση κινδύνου και τους εκπρόσωπους της διαχείρισης αυτής θα πρέπει να διευκρινιστεί και να ενισχυθεί. Ε, με υπέρ ενός νομοθετικού πλαισίου στην ε, εταιρική διακυβέρνηση. Θα λάβει χώρα, χώρα διάλογος με όλους τους εμπλεκομένους, ε, γιατί αυτό είναι σημαντικό σήμα που θα δώσουμε στους πολίτες μας, ότι όντως έχουμε σοβαρά την πρόθεση να ε, εισαγάγουμε υγιείς κανόνες στην οικονομία. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνεται η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12 για τις διεκθέσεις. Ευχαριστώ τους συναδέλφους, ευχαριστώ και τον Επίτροπο. Και μπορούμε να περάσουμε στην ώρα των ερωτήσεων.